Okay, we are already delayed a little bit. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τη συνεδρίασή μας. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σημείο 19 για την ε, η ερευνητική συνάντηση στη Σουηδία. Αυτό έχει αναβληθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο ότι αντιστρέφονται τα σημεία 7 και 8. Πρώτα δηλαδή θα συζητήσουμε το 8 και μετά το 7 κατόπιν επιθυμίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να τους ευκολύνουμε. Σημείο 3 δεν έχουμε πρακτικά προσέγγιση. Προχωράμε στο σημείο 4. Λείπαμε λίγο που σας ενημερώνω ότι ένα από τα μέλη του προσωπικού μας που ήταν μαζί μας πολύ καιρό, η Ζορζάνα Σάντου, έχει ε, αποχωρήσει από τη γραμματεία. Είναι εδώ σήμερα. Ε, έχετε πάρει στη γραμματεία της ΦΑΜ. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που σας χάνουμε εμείς. Συγχαίρω την γραμματεία της ΦΑΜ που ε, σας κέρδισε. Σας εύχομαι ε, ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Τζορτζιάννα, για όλη τη δουλειά που έχει κάνει για την Επιτροπή μας και για την ευγένειά σου. να πάντα θετική και ευγενική απέναντι σε όλους. Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Άλλη μία ανακοίνωση έχω. Έχουμε δύο ασκούμενους στην γραμματεία. Έλεν ράχε και Αλεσάνδρο Κρανάτο. Πού βρίσκεστε? Πίσω, πίσω. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εύχομαι να περάσετε πολύ καλά στην γραμματεία ως ασκούμενη. Αν ε, είναι κανείς αυστηρός μαζί σας, πάρτε με τηλέφωνο. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί σας. Δεν έχουμε παρατηρήσει για το σημείο 5 που είναι τα διάφορα. Οπότε περνάμε στην ε, παρουσίαση της ε, έκθεσης ε, για το 2017 για τους πολίτες, ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών. Και χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω την Τίνα Άστολα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενικής Διευθύντριας για τη Δικαιοσύνη και τους Καταναλωτές. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σε λίγες μέρες ε, θα γιορτάσουμε την 60η επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης. Ε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας κοινό χώρος ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και είναι κατάλληλη στιγμή να υποβάλουμε την ε, έκθεση ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, για το 2017 που υιοθέτησε στις 24 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ευρωπαϊκή υπηκότητα, η ηθαγένεια, δεν ε, αντικαθιστά, προστίθεται στην εθνική υπηκότητα και την εκτιμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες διότι συνδέεται με θεμελιώδη δικαιώματα και προνόμια. Έχει να κάνει και με κοινέ αξίες που ενώνουν Εμά τους Ευρωπαίους. Όπως επιβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ηθαγένεια της ε, Ένωσης ε, θα πρέπει να είναι το θεμελιώδες καθεστώς των ε, υπηκών των κρατών μελών. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι ακρογωνία λήθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να είναι για τους πολίτες ό,τι είναι και το ευρώ για την ΟΝΕ. Είναι ακόμα πιο σημαντικό στο ισχύον πολιτικό πλαίσιο να αναλάβουμε την ευθύνη και να αναλάβουμε τα απαραίτητα βήματα για ε, προς όφελος των πολιτών της, Ευρω... της Ευρώπης. Όσον αφορά την έκθεση, το άρθρο 25 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τρία χρόνια να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την ΕΟΚΕ σχετικά με την εφαρμογή των ε, διατάξεων της συνθήκης ε, σχετικά με την ηθαγένεια και, την, ε, και τις μη διακρίσεις. Τρίτη φορά λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μία δέσμη δύο εκθέσεων. Την έκθεση για την ηθαγένεια, ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μία ένωση δημοκρατικών αλλαγών που κοιτάει το μέλλον και την έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2013 στο 2016 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων ε, για μη διάκριση και ηθαγένεια στην Ένωση. Και οι δύο αυτές εκθέσεις έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Έχουμε επίσης ε, εκδώσει ενημερωτικά δελτία που συνοψίζουν τα βασικά σημεία των εκθέσεων αυτών σε όλες τις γλώσσες και συνεχίζεται η διάδοση των εκθέσεων αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έκθεση του 2017, η δέσμη μάλλον αυτή των εκθέσεων, ε, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σύμφωνα με τις πολιτικές της προτεραιότητες και τις επιτρέπει επίσης να θεσπίσει προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά του τομεί προτεραιότητας, πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ήδη έχουμε πετύχει πολλά. Το 87% των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι εκτός από την ηθαγένεια τους στο κράτος μέλος, ότι είναι και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Για να μπορέσουν ε, να εκμεταλλευτούν ε, στο έπακρον ε, τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά και πώς μπορούν ε, να τα ασκήσουν. Για παράδειγμα, το δικαίωμα προξενικής προστασίας ε, είναι κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν πολλά ακόμα οι πολίτες. Και δεν γνωρίζουν τι επίπεδο προστασίας τους προσφέρεται. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε στους πολίτες να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους αυτά και να μπορέσουν να τα ασκήσουν. Πολλοί Ευρωπαίοι επίσης ε, δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι σημαντικό να ψηφίζουν στις ευρωεκλογέ. Πολλοί δεν έχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν όταν ε, δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή, Ένωση θα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ώστε οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν καλύτερα το περιεχόμενο ε, και τη σημασία των δικαιωμάτων τους ως ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει προξενικά δικαιώματα ε, και εκλογικά δικαιώματα. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με διάφορους ενδιαφερόμενους κύκλους συμπεριλαμβανομένων τοπικών και περιφερειακών αρχών ώστε να φροντίσουμε οι πολίτες να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Όσον αφορά τον δεύτερο τομέα προτεραιότητα, θέλουμε να ενθαρρύνουμε του πολίτε να συμμετέχουν ενεργά στην ε, δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι δεν ασκούν ε, πλήρως ε, τα δημοκρατικά και εκλογικά τους δικαιώματα το 42% είναι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και αυτό είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτοί που ψηφίζουν πρώτη φορά είναι η μεγαλύτερη ομάδα αυτών που απήχαν στις τελευταίες εκλογές. Ταυτόχρονα οι νέοι ενδιαφέρονται πολύ να συζητήσουν πολιτικά θέματα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ε, αυτά τα πράγματα δεν φαίνεται να ταιριάζουν καλά μεταξύ τους ε, και αυτό είναι πρόβλημα. Στην υπηρεσία μας 8 στους 10 λένε ότι θα ασκούσαν πλήρως τα δικαιώματά τους αν γνώριζαν καλύτερα τα ωφέλη. Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν τα περί των ευρωεκλογών και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή. Θα πρέπει να γνωρίζουν τι διακυβεύεται όταν δεν ψηφίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για την παροχή των σχετικών πληροφοριών. Θα έχουμε διαλόγους με τους πολίτες για να ενθαρρύνουμε δημόσιο διάλογο και να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Θα προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να ψηφίσουν και να θέσουν και υποψηφιότητα σε ευρωεκλογέ το 2019. Και του χρόνου θα οργανώσουμε μία εκδήλωση υψηλού επίπεδου για την δημοκρατική συμμετοχή και θα δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές ε, για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ε, των νέων και άλλων ομάδων που δεν ε, εκπροσωπούνται επαρκώς. Τρίτος τομέας προτεραιότητας. Θα θέλουμε να απλοποιήσουμε την καθημερινή ζωή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας μαζί με την ειρήνη είναι τα δύο πιο σημαντικά επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών και αυτά που εκτιμώνται περισσότερο. Το να μπορεί κανείς να ταξιδεύει, να σπουδάζει, να εργάζεται και να διαμένει σε άλλα κράτη-μέλη είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες. 7 στους 10 πιστεύουν ότι η ελευθερία ε, κυκλοφορίας ε, είναι ε, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όχι μόνο για αυτού, αλλά και για την οικονομία της χώρας τους. Το 56% θεωρούν ότι αυτή η ελευθερία είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, η ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε προσπάθειες ε, για να διασφαλίσει την ε, επιβολή της νομοθεσίας ε, που έχει οδηγήσει σε μεταφορά τις οδηγίες για την ελεύθερη κυκλοφορία στο δίκαιο των περισσότερων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση για να διασφαλίσει την ε, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχει η έκθεση πρωτοβουλίας της ΠΕΤΗ και της ΛΥΜΠΕ για τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία. Θα... Ε, όπου διαπιστώνεται το τι θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουν οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, ακολουθήσει τις συστάσεις, ε, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των πολιτών ε, και των συγγενών τους σχετικά με τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Όλα αυτά αποτελούν κοινή ευθύνη, τα οποία θα πρέπει να πετύχουμε με κοινέ προσπάθειες. Το να διαμένει ε, κανείς σε άλλο κράτος μέλος ε, συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση. Πολλοί από εμάς το γνωρίζουμε αυτό. Πολλοί πολίτες ε, διαπιστώνουν ε, ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι, διαρκούν πολύ, ότι είναι δύσκολες οι διασυνοριακές υποθέσεις. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δημιουργήσει μία ενιαία δικτυακή πύλη που θα συνδέει πληροφορίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι πολίτες να έχουν εύκολη επιγραμμική πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστήριξη, ιδιαίτερα όταν μετακομίζουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Μαζί με την ε, έκθεση η για το 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ξεκινήσει ε, τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου που στόχο έχει να διασφαλίσει οι Ευρωπαίοι πολίτες όπου και να βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, συνομιλούν με ε, ε, αξιωματούχους υπαλλήλους που να γνωρίζουν απολύτως τα δικαιώματά τους και να μπορούν να τους βοηθήσουν να τα ασκήσουν. Τέλος, θέλουμε να προωθήσουμε την ισότητα και να είναι οι πολίτες μας ασφαλείς. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση και ελευθερία ε, για να απολαύουν ελεύθερα των δικαιωμάτων τους. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συγγενείς τους μπορούν ε, να ε, συναντήσουν δυσκολίες κατά την χρήση της, της ταυτότητάς τους ή άλλων εγγράφων. Κάποια έγγραφα είναι πολύ λιγότερο ασφαλή από άλλα. Και όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους να βελτιωθεί η ασφάλεια των δελτίων ε, ταυτότητας και αδειών παραμονής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, συγγενών τους ε, από τρίτες χώρες. Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση εις βάρος κανενός ε, λόγω φύλου, ε, καταγωγής, ε, θρησκείας ή για άλλο λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει εκστρατεία για να καταπολεμηθεί η βία εις βάρος των γυναικών με συγκεκριμένες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης, στηρίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, για την πρόληψη της βίας εις βάρος των γυναικών. Θα συνεχίσουμε επίσης ε, να στηρίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, σχετικά με την οδηγία κατά των διακρίσεων, καθώς επίσης και το θέμα των ατόμων ΛΟΑΔ. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Πιστεύω ότι τον επικεντρωθούμε σε αυτούς τους τέσσερις τομείς με την υποστήριξή σας. Ε, σημαίνει ότι οι πολίτες μας θα μπορέσουν να απολάβουν πλήρως των δικαιωμάτων τους χωρίς διακρίσεις ε, ε, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι βέβαιο ότι η εκπόνηση, η διαμόρφωση αυτού του θεματολογίου δεν ε, αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί συλλογική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και φυσικά σημαντικό ρόλο έχει να παίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Άστολα. Το θωρώ εντελώς αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι 87% των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν πολύ καλά τα δικαιώματά τους. Μας το επισημάνατε και χαίρομαι ιδιαίτερως. Η προτεραιότητά σας είναι εξαιρετική. Οι πολίτες διαμορφώνουν ε, ε, τα θέματα αυτής της Επιτροπής κάθε χρόνο και αυτό επιβεβαιώνεται στις αιτήσεις εκθέσεις για τις αναφορές ε, σε, στις εκθέσεις για την αιτήσια δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών. Θα ετοιμάσουμε την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση για την Ιθαγένεια και θα έχουμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας σε συνεργασία με την Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών και βάσει του κανόνα 54. Η κυρία Μπεσέρα θα είναι η συγγήτρια. Τώρα, δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κυρία Τανούκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα όχι μόνο για να μιλήσουμε για τις τρέχουσες υποθέσεις μας, αλλά για να προχωρήσουμε και με τις νέες προτάσεις για την Ιθαγένεια. Προς το παρόν, έχει γίνει μια συζήτηση για την ελευθερία της μετακίνησης, αλλά αυτό είναι μόνο μία από τις διαστάσεις της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. είναι κάτι που απορρέει από το, την ηθαγένεια κράτους μέλους. Δηλαδή κάποιος έχει την ευρωπαϊκή ηθαγένεια επειδή έχει την ηθαγένεια συγκεκριμένου κράτους μέλους. Υπήρχε μια επιλογή να δοθεί και στους μονίμως διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς μέρος του Κοινοβουλίου αντιστάθηκε σε αυτό. Για παράδειγμα, η έκθεσή μου δεν προχώρησε στην αντίστοιχη επιτροπή. Με το Brexit όλο και περισσότεροι άνθρωποι και περισσότεροι πολιτικοί συνειδητοποίησαν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, τι σημαίνει και πώς μπορεί να δοθούν δικαιώματα σε Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στα κράτη-μέλη. Και υπάρχει και το πρόβλημα των απάτριδων στην Λετωνία και στην Εσθονία. Οι μόνιμοι διαμένοντες έχουν την προστασία των κρατών, έχουν διαβατήρια που εκδίδονται από τα κρατημέλη, έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό για τις θεωρήσεις. Θα ήταν φυσικό να έχουν και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την επέκταση των δικαιωμάτων και σε μη ε, ε, σε πολίτες που δεν έχουν ηθαγένεια κάποιου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ε, καλυφθούν και όσοι είναι μόνιμος, μονίμως διαμένοντες και δεν είναι υπήκοοι χώρας. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Ο Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της έκθεσής της. Εάν δει κανείς ε, τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Brexit, ίσως η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να εξεταστεί. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια θα πρέπει να ενισχύει το αίσθημα, την αίσθηση της αλληλεγγύης και σε τάση φιλοευρωπαϊκή από πλευράς πολιτών. καλό θα είναι να γίνει μια εξτρατεία ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για το ποια είναι τα δικαιώματά τους και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αναλάβουν τα δικαιώματά τους, να τα ασκούν και θα πρέπει να γίνει και πολιτική συζήτηση. Η θαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το να είναι κανείς πολίτης ενός κράτους μέλους. Επειδή είμαι υπηκό συγκεκριμένη χώρα που είναι μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα πρέπει να μην την υποβαθμίσουμε. Γιατί τελείως δεν θα έχει νόημα και πολύ νόημα. Εάν τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έφυγε, έφυγαν. Άρα, ή στι διαπραγματεύσει θα βρούμε κάποιο καθεστώς για αυτού του πολίτε που είναι διαμένοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα έχουν το ίδιο καθεστώ με του Καναδού, για παράδειγμα. Μιλώ για του Βρετανού που μένουν στι υπόλοιπε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση για να δούμε πώ θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι θέμα προσυζήτηση πράγματι. Εάν τώρα η έκθεση λέει ότι οι πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα ασκούν, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι καλή αλλαγή. Εμείς πάντοτε ξεκινήσαμε από κάτω, από τη βάση της πυραμίδας για να προχωρήσουμε προς τα πάνω και αυτό είναι ακριβώς αυτό που ε, ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι εξ ονόματος της Μπέατρίθ. Δεν θα το διαβάσω βέβαια, γιατί ίσως ε, έρθει και μιλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κάποια αντίφαση. Νόμιζα ότι η συζήτηση είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μιλώ για συγκεκριμένο διαβατήριο πράσινο ή γκρι, συγκεκριμένου χρώματος. Ίσως έχει σχέση με τη διατύπωση σε κάποιες γλώσσες. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι κάτι το πιο ευρύ, κάτι το πιο πνευματικό, πιο αφηρημένο θα έλεγα, διανοητικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα μεταξύ των διαφόρων συνομιλητών. Ε, υπάρχει κάποιος που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, πέντε χρόνια και δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει στις ευρωεκλογές. Είναι καλή έκθεση θα είπα ότι θα τη διαβάσω και τελικά πέρασα δύο-τρεις ώρες και ξενύχτασα διαβάζοντάς τη. Εν πάση περιπτώσει η έκθεση είναι καλή, ε, δίνει λαβή για μια επικοδομητική συζήτηση και ελπίζω να βρούμε λύσεις ε, σε αυτά τα σημεία στα οποία έχει σημειωθεί τέλμα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά δίνω το λόγο στην κυρία Άστολα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, έχω πράγματα να πω που θα σας εκπλήξουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ακολουθεί την Ιθαγένεια των κρατών μελών. Ως προς το Brexit, Δεν λέμε κάτι για τις διαπραγματεύσεις, δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, θα ξεκινήσουν λίγαν συντόμως. Θα λάβουμε την επιστολή κοινοποίησης. Δεν θα ήθελα να αρχίσω να μαντεύω ποια μπορεί να είναι η κατάσταση των υπηκών του Ηνωμένου Βασιλείου αργότερα. Θα είναι υπήκοοι τρίτων χωρών εάν δεν γίνει διαπραγμάτευση για κάποιο άλλο καθεστώς για αυτούς. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, να εφιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι εμείς μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΑ θα οργανώσουμε μία συζήτηση, ακρόαση, στις 29 Ιουνίου για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, άρα πριν επέλθει το Brexit, όχι, 4 Μαΐου, συγγνώμη, με διορθώνουν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να, λάβουμε, να θεωρήσουμε δεδομένο το γεγονός ότι 3,1 Ευρωπαίοι πολίτες μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 2 εκατομμύρια Βρετανοί πολίτες μένουν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες των λοιπόν χωρών μελών μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως. Και αυτό το θέμα τους αφορά. Είμαι σε συνεχή διάλογο με τον Μισελ Μπαγνιέ, τον πρώην Επίτροπο και ε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τον Brexit ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέστησε σαφές ότι θα θέσει τους πολίτες πολύ ψηλά, στη πιο ψηλή θέση στο κατάλογο των προτεραιοτήτων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο παρακαλώ με το θέμα αυτό. Αυτή είναι η ακρόαση για τους απάτριδες. Η ακρόαση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στις 4 Μαΐου. Σας ευχαριστώ κύριε Άστολε που ήρθατε, που μας παρουσιάσατε την έκθεση. Πράγματι τα, όλα είναι ρόδινα στην πραγματική ζωή. Θα το διαβάσω όλο αυτό το κείμενο πολύ προσεκτικά. Τώρα ε, καλώ τον κύριο Παλσάτη να προεδρεύσει για το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι ένα θέμα που αφορά την Ισπανία. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα αποχωρήσω από την αίθουσα. Εν τω μεταξύ θα συνεχίσετε με άλλη προεδρεύουσα, με άλλο προεδρεύοντα. Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, magyar nyelvet fogom használni. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Καλή σας μέρα. Θα μιλήσω ουγγρικά στη διάρκεια της Προεδρίας μου. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εξέταση της αναφοράς 0043 κάθετος 2004 της ε, Άννα Ρίτα Αμορόζο, η οποία αν θυμάμαι καλά ε, βρίσκεται μεταξύ μας. Πρόκειται για μία αναφορά η οποία η οποία ε, αφορά τα διόδια αυτοκινητοδρόμων που έχει επιβάλει η Γερμανία στους δικούς της αυτοκινητοδρόμους. Αυτό θα συζητήσουμε, αυτό είναι το θέμα μας το ε, σημερινό και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, αναφέρουσα, την κυρία Άννα Ρίτα Αμορόζο. Gentile Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, στις 15 Μαρτίου τρέχοντος έτους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ε, ενέκρινε το ψήφισμα της ε, κυρίας Καριμάντελη εξ ονόματος Επιτροπής Τουρισμού και Μεταφορών σε απάντηση της προφορικής απάντησης της Επιτρόπου Βελέτα Μπούλτς σχετικά με την υπόθεση της Γερμανίας η οποία προτίθεται να χρεώσει διόδια μονάχα στους ξένους που κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους της ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία τα οποία ε, όμως ε, αποτελούν παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της μη διακριτικής μεταχείρισης έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 18 τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω υπογράψει αυτήν την αναφορά αλλά ακόμα σήμερα παραμένω ε, χωρίς ε, ε, συγκεκριμένη απάντηση όσον αφορά την κατάργηση αυτού του συστήματος διοδίων που βασίζεται στην ε, εθνικότητα και που επομένως ε, παρεμποδίζει την διαμεθοριακή κινητικότητα. Ε, μία κρυμμένη διακριτική μεταχείριση η οποία εξακολουθεί να υφίσταται έστω ως υποψία ακόμα και αν έχει αρθεί η διαδικασία επί παραβάση. Και θεωρούμε ότι το στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε, ότι αναφέρθηκε μονάχα ως προεκλογικό ε, πρόγραμμα δεν μας πείθει. Το θέμα των μεταφορών αντιπροσωπεύει έναν από τους ε, ε, τομείς κοινή πολιτικής εδώ και 30 χρόνια και επιπλέον. Το άνοιγμα λοιπόν της αγοράς των μεταφορών είναι ουσιώδου σημασίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ε, ε, ανταγωνισμού σωστού ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και μάλιστα χωρίς επιπλέον κόστος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει αναφερθεί σε ψηφίσματά του κατά την έννοια αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν επίσης έχει παρέμβει λέγοντας ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εισάγουν ε, διακριτικά συστήματα ε, ε, διοδίων. Συγκεκριμένα, το 1996 παρενέβη όσον αφορά το σύστημα βινιέτας, δηλαδή σήματος για αυτοκίνητα διαρκείας μίας εβδομάδας στην Αυστρία, έτσι ώστε να μην υπάρξει διακριτική μεταχείριση των τουριστών. Επίσης, το 2014, όταν η Σλοβενία εισήγαγε ένα σύστημα σήματος βινιέτας για τους ξένους, του οποίου η τιμή ήταν αναλογική λογική με το σύστημα ε, των ε, μακροχρόνιων σημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι, ε, πολύ και διάφοροι, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διάκριση ε, όσον αφορά την πληρωμή διοδίων στα κράτη-μέλη. Μπορεί κανείς να αναφερθεί στην αρχή του όποιο μολύνει πληρώνει, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να πληρώνονται τα διόδια ε, και να έχουν κόστο ανάλογο με την διαδρομή και επομένω να μην υπάρχει καμία συσχέτιση με το τέλος κυκλοφορίας το οποίο πληρώνουν όλοι. Η αρχή του όποιος μολύνει πληρώνει ε, έχει αποτελέσει επομένως βάση του συστήματος της ευρωβινιέτας, του ευρωσήματος. Ε, όμως αγνοήθηκε στην περίπτωση της γερμανικής ε, πρότασης γιατί στην προκείμενη περίπτωση θεωρείται ότι η δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη να επανα τα και να επανεπενδύσουν τα χρήματα ε, σε συγκεκριμένες υποδομές υψηλού ευρωπαϊκού ε, ε, ευρωπαϊκής σημασίας αυτή η διασύνδεση λέω δεν αναγνωρίζεται η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης βάσει της εθνικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ως αρχή με αυτήν της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα δικαίωμα επομένως το οποίο θα πρέπει περαιτέρω ενδιαφέρον να ενισχυθεί ε, μέσω της ε, ενίσχυσης ε, της αίσθησης του ανήκεινε σε μια κοινότητα. Το άρθρο 21 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ότι η αρχή της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει άμεση ισχύ και δίνει στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα για ίδια νομική άσκηση του δικαιώματός του της ελεύθερης κυκλοφορίας και της διαμονής. Δεν κάνει όμως καμία αναφορά σε οικονομικό συσχετισμό σε σχέση με την δραστηριότητά του. Εγώ ζητώ από την, Επιτροπή Αναφορών να γίνει δεκτή και να, παρα... Ε, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μου και να ζητηθεί η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ως θεματοφύλακα και προστάτητα των συνθήκων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και επομένως να ε, αρθεί οποιαδήποτε υποψία και επομένως ε, να μπορέσει να, ε, της άρσης της διαδικασίας επιπαραβάση και να μπορέσει η Γερμανία να φτάσει ενώπιον των δικαστηρίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Is Mr. Peter Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητή κυρία, καλημέρα σας. Με λένε Πίτερ Ντεμέγερ και ε, εργάζομαι στο τμήμα συντονισμού της DG Move και μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τη θέση μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πράγματι η υπόθεση αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ένας πολύ σημαντικός ε, φάκελος στην παρέμβασή σας αναφέρετε και καλώς ότι η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει είναι ε, βασική αρχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιθυμεί να εφαρμόζεται παντού. Να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπατε. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε εμείς την κατάσταση είναι η κα... Είναι ο εξής. Όταν η Γερμανία προσπαθεί να επιβάλλει ε, διόδια ε, στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους με ε, την, το κόλλημα ενός αυτοκόλλητου στο παρμπρίζ που δείχνει ότι έχει υπάρξει πληρωμή. Αυτό ισχύει για όλους τους χρήστες, ε, Γερμανούς πολίτες και μη. Υπάρχει πλήρης διάλογος με τις γερμανικές αρχές, πολλά έχει πει ο τύπος, αλλά μέχρι ότου υιοθετήσει το Γερμανικό Κοινοβούλιο το νομοθέτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει ε, τα προσχέδια της νομοθεσίας. Σημειώνουμε τα περιεχόμενα του φακέλου, αλλά πρέπει να περιμένουμε να νομοθετήσει οριστικά το Γερμανικό Κοινοβούλιο για να αποφανθούμε. Όλα αυτά αποτελούν ε, μέρος του πακέτου νομοθετικών προτάσεων που ε, προετοιμάζουμε ε, κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου και δεν είναι καθόλου σαφές σε ποιο βαθμό η νέα πρόταση θα ισχύσει και για τα επιβατικά οχήματα, αλλά κατά τη διάρκεια του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση νομοθετικού πακέτου για την επιβολή για την χρήση των δρόμων, αλλά και για τις ε, οδικές μεταφορές και ε, τέτοια θέματα θα εξεταστούν. Σε αυτό το πλαίσιο ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής η θέση. Ο Πίτερ. Ναι. Ε, και εγώ νομίζω ότι δεν είναι αδικαιολόγητη η θέση της αναφέρουσας. Η Κομισιόν βρίσκεται σε διάλογο με τις εθνικές αρχές. Δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν τέτοια μέτρα σε διακρίσεις και, και εγώ Γερμανός είμαι. Και από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με ε, την ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ε, ο διάλογος αυτός συνεχίζεται. Έχουν αρκετά θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Προτείνω λοιπόν, εφόσον δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου ε, να περάσει το θέμα από το Γερμανικό ε, Κοινοβούλιο και να δούμε ακριβώς πώς έχει η νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος ευρωβουλευτής που να θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Αμορόζο. Ακούσαμε την αναφορά σας, ακούσαμε τις προτάσει των συναδέλφων. Θα αφήσουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά αυτή και θα περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε από τις ε, Εθνικές Αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνείτε? Ωραία. Κυρίες και κύριοι, Περνάμε στην αναφορά 2334 του 2014. Ο Ισπανός υπήκος, ο κύριος Πορτέλα, έχει υποβάλει αυτή την αναφορά σχετικά με θέματα φορολογίας. Πέντε λεπτά έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνομαι στην Επιτροπή Αναφορών εξ ονόματος της Εθνικής Συντονίστριας των μεταναστών που έχουν επιστρέψει στη Γαλλικία. Είναι ένα συντονιστικό όργανο που εκπροσωπεί χιλιάδες ε, Γαλλικιανούς συνταξιούχους που αντί να απολαμβάνουν τη σύνταξή τους είναι υποχρεωμένοι να βγαίνουν στον δρόμο για να διαδηλώνουν γιατί υφίστανται τη φορολογική παρενόχληση και επίθεση της Ισπανικής εφορίας. Είναι ένα σύλλογο μεταναστών Ισπανών που πέρασαν τη ζωή τους εργαζόμενοι στο εξωτερικό ως μετανάστες. Θεώρησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος όπου δεν θα υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ κρατών μελών και θα είναι ένας κοινό χώρος δικαιωμάτων. Πλήττονται λοιπόν από το Ισπανικό κράτος σε μεγάλο βάθος. Ο αναφέρον σε σχέση με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 25 Νοεμβρίου του 2015 θεωρεί ότι η Ισπανική κυβέρνηση επιβάλλει ε, διακρισιακή και διακριτική φορολόγηση, κάνει διακρίσεις σε φορολογικό επίπεδο. Γιατί οι, οι Ισπανοί μετανάστες έχουν ε, συντάξεις από άλλες χώρες και τους υποχρεώνει η Ισπανία να ε, πληρώσουν φόρα γι' αυτό σε σχέση με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δεν συμφωνεί με την άποψη αυτή, πρέπει να πούμε ότι Προφανώς ο, ο κάθε Ισπανός συνταξιούχος μπορεί να προσφύγει στην Ισπανική δικαιοσύνη. Όμως αυτό το οποίο λέει ο αναφέρον είναι ότι έτσι θα αποφευχθούν τα τεράστια προβλήματα των συνταξιούχων μεταναστών που επέστρεψαν στη χώρα τους και που μένουν σε μεγάλο βαθμό στην Ήπεθρο και που δεν έχουν πολλές δυνατότητες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Είναι ένα συλλογικό πρόβλημα το οποίο λύνουν ε, ατομικά τα ισπανικά δικαστήρια προς όφελος του καθενός. Δηλαδή κάθε ένας συνταξιούχος που λαμβάνει γερμανική σύνταξη ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Ε, κάθε ένας από αυτούς τους χιλιάδες, ενώ έχουμε διάφορες αποφάσεις ισπανικών δικαστηρίων προς όφελος άλλου αντίστοιχου που έχει υποστεί το ίδιο, μιλούμε για 13.000 ανθρώπους. Κάποιοι έχουν διεκαιωθεί στα δικαστήρια. Πρέπει να πάνε όλοι και να δικαιωθούν. Γι' αυτό θα έπρεπε η Επιτροπή Αναφορών να αποβαθεί προ όφελό του και να μην περιμένει και να περιορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να του προτείνει να προσφύγουν στην Ισπανική δικαιοσύνη. Και γι' αυτό ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μα. Ε, για όσο χρόνο ε, ε, συνεχίζει και παρατείνεται και παραμένει αυτή η φορολογική επίθεση του Ισπανικού κράτους σε βάρος ε, συνταξιούχων της Γαλλικίας. Ε, η Γαλλικιανία είναι ένας λαός που ανέκαθεν μετανάστευε και ανέκαθεν με ταξίδευε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χουάν Λόπεθ Ροδρίγες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος ε, της ε, Ταξούντ και θα απαντήσω σε σχέση με την αναφορά του κυρίου Λαγοπορτέλα. Ε, βεβαίως εμείς ε, με μεγάλη ευαισθησία ε, στεκόμαστε στο ζήτημα των συνταξιούχων που προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους και τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν στις δικαστικές διαδικασίες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν, αυτά θα πρέπει να λυθούν σε σχέση με την συμφωνία που η χώρα, η Ισπανία, έχει υπογράψει με άλλε χώρες. Πρόκειται για, μια, για ένα πεδίο το οποίο δεν έχει εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. και επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάρει θέση. Επίσης, όσον αφορά ε, τις συντάξεις αναπηρίας, επίσης και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει εναρμονισμένη ε, νομοθεσία όσον αφορά τις συντάξεις ε, αναπηρίας και επομένως έχει δικαίωμα η Ισπανία να ζητήσει εξακρίβωση του βαθμού αναπηρίας. Επίσης, ε, πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία αποφασίζει ε, για το κατά πόσον αυτές οι συντάξεις αναπηρίας θα εξαιρούνται φόρου ανεξάρτητα από το ποια είναι η χώρα στην οποία έχει εκδοθεί και που πληρώνει τη σύνταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο σε όποιον το ζητάει. Η Ρόζα παρακαλώ. Ρόζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω τον αναφέροντα και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Το πρόβλημα ε, προκύπτει γιατί υπάρχουν κάποιες ε, φορολογικές δυσκολίες, ε, γιατί προκύπτει δυσκολία για περίπτωση αναπηρίας, ειδικά όταν τη σύνταξη δεν την δίνει το ισπανικό σύστημα, αλλά κάποιο άλλο. Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι υπεύθυνα για τέτοια ζητήματα γιατί δεν υπάρχει εναρμόνιση και επομένως αυτό το θέμα αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Ωστόσο, να δούμε λίγο τι έκανε η Ισπανική κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση της Γαλλικίας ασχολήθηκε με το θέμα από την αρχή και είπε ότι ε, η φορολόγηση των μεταναστών ε, τους απασχολούσε πάρα πολύ. Ε, έγιναν διάφορες συνεδριάσεις με τους ενδιαφερόμενους. Νεύουν αρνητικά οι αναφέροντες. Όχι, όχι, εγώ έχω τις ημερομηνίες στις οποίες συνεδρίασε η Τζούντα της Γαλλικίας με το θέμα αυτό. Ε, μέσω ε, λοιπόν και της κυβέρνησης της Γαλλικίας ξεκίνησε και μία ε, εκστρατεία με επιστολές προς την κεντρική κυβέρνηση. Αναφερθήκατε μάλιστα, ο αναφέρον έθιξε και το ζήτημα αυτό. Και επίσης ο επικεφαλής της κυβέρνησης ε, της ε, ε, Γαλλικίας ήρθε σε επαφή επανειλημμένα με τον αρμόδιο υπουργό του κ. Μοντόρο και ακριβώς ζήτησε από τον υπουργό και από το Υπουργείο να σκύψει πάνω στο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την κατάσταση. Τέλος, σε σχέση με όλα αυτά πρέπει να πω ότι ως αποτέλεσμα των ε, προσπαθειών ε, της ε, κυβέρνησης της Γαλλικίας έχει υποβληθεί τροπολογία στη φορολογία, στην νομοθέτηση της φορολογίας εισοδήματος ε, και ε, το 2015 δόθηκε εξάμηνη παράτηση για την διευθέτηση ε, όλων των κυρώσεων των ενδιαφερομένων αυτών ανθρώπων χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση λόγω τόκων. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, συμφωνώ με την ε, Κομισιόν ότι εδώ μιλάμε για αρμοδιότητα ε, της ε, Ισπανικής κυβέρνησης και η τοπική κυβέρνηση της Γαλλικίας σωστά προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να λύσει το θέμα. Εγώ θα, θα ήθελα να μπορούσα να σας δώσω μια άλλη απάντηση, δηλαδή ότι είμαστε αρμόδιοι για το θέμα και επομένως μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Ε, είναι γεγονό ότι μερικές φορές προκύπτουν προσδοκίες στα πλαίσια της Επιτροπής μας αναφορών για θέματα που όμως δυστυχώ δεν αποτελούν αρμοδιότητά μας. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι και αντιπρόεδρος ε, της ε, ομάδας για την αναπηρία και είναι γεγονός ότι εάν κάποιος είναι ε, δηλωμένος και αναγνωρισμένος ως ανάπηρος στην Ισπανία, δεν μπορεί με το ίδιο αυτό χαρτί να πάει στη Γερμανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και να ζητήσει εξαίρεση φόρου ή οτιδήποτε ε, άλλο. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους ε, εναρμόνιση όσον αφορά τα θέματα αυτά, γιατί δεν έχει ε, έννοια. Ε, αυτό, αυτή η διαδικασία και αυτή η κατάσταση απλώς προκαλεί τρομερά προσκόμματα, εμπόδια σε όλη την Ευρώπη και είναι παράλογο. Ωστόσο η κατάσταση σήμερα έχει ως έχει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθες ξεκίνησε τη λειτουργία του το δίκτυο για τις αναφορές. Και φαντάζομαι ότι ετούτη η αναφορά θα μπορούσε να εξεταστεί υπό αυτό το φως. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αναφορών. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτό και δεν μπορούμε να απογοητεύουμε τους αναφέροντες λέγοντας ότι αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της, του Ισπανικού κράτους. Νομίζω ότι σαφώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και η κυρία Σάββας Φερακούτα αναφέρθηκε ε, στην θέση αυτή των ατόμων με αναπηρίες. Που διαφέρει μάλιστα ανάλογα με το κράτος μέλος. Η πρότασή μου είναι να στείλουμε αυτή την αναφορά στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, που συμμετέχει επίσης στο δίκτυο. Ως μέλος της Επιτροπής αυτής ε, μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναφορά αυτή. Ιδιαίτερα καθότι η η εφαρμογή του θεματολογίου για τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελεί ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση Juncker. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όσον αφορά τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, και να τη στείλουμε προς ενημέρωση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είναι θλιβερό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που λέει σε αυτό το σύλλογο συνταξιούχων που έρχεται εδώ αναζητώντας δικαιοσύνη είναι να τους λέει ότι έχουν δικαίωμα να πάνε στα δικαστήρια. Μα το ξέραν αυτό ούτως ή άλλως. Δεν ήρθαν εδώ για να τους πούμε να πάνε στα δικαστήρια. Επίσης θλιβερό, θλιβερή είναι η διγλωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χθες, για άλλο ζήτημα που είχε να κάνει με τις συντάξεις και την Νορβηγία, μιλούσαμε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μας είπε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί η Νορβηγία δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όμως που η Ισπανία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε να πάει στα δικαστήρια. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει περισσότερα, μπορεί να κάνει έτσι ώστε αυτή η κατάσταση αδικίας και διακρίσεων που επιβάλλει η Ισπανική κυβέρνηση και το Ισπανικό κράτος να λυθεί ως πρόβλημα. Αυτά τα δύο είναι θλιβερά. Κατά τρίτο λόγο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Πρέπει να αναλάβουμε τις προτάσεις των αναφέροντων να θεωρήσουμε υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Καταρχάς, μια ερώτηση. Ο πω και έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και ρωτάει αν η νομική υπηρεσία θα μπορούσε να πάρει θέση στο θέμα αυτό, εάν είναι σωστή δηλαδή αυτή η νομική αντίληψη του θέματος. Επίσης, μια δική μου εκτίμηση. Μια, μια δική μου εκτίμηση. Αυτό έχει να κάνει με το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ανθρώπους που να μεγαλώνουν σε ένα κράτος μέλος, να ζουν σε άλλο, να, ενδεχομένως να λαμβάνουν τη σύνταξή τους σε τρίτο κράτος μέλος. Έτσι είναι η ζωή. Ας Φανταστούμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και ε, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Να μην ε, αναγνωρίζεται, για παράδειγμα, το καθεστώς τους σε άλλο κράτος μέλος. Και να έχουμε περιπτώσεις εκ των υστέρων φορολόγησης. Δεν είναι ωραίο αυτό. το πρόβλημα και μήπως να υπερασπιστούμε και το λίγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι είναι θέμα αρμοδιοτήτων. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ε, κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι με το μέρος των αναφερόντων. Ε, θα έλεγα, μα, αγαπητά κράτη-μέλη, ε, να θίξετε το θέμα, να το θέσετε επιτάπητος και να βρείτε μια λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά να το επιβεβαιώσω αυτή είναι η νομική υπηρεσία, νομίζω ότι είναι ο λάθος συνομιλητής, διότι δεν έχει την σχετική αρμοδιότητα. Ε, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ωραία δεν είναι αρμόδια να κλείσουμε την αναφορά, το πρόβλημα όμως παραμένει. Μήπως να παραπευθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή ναι, είναι άδικο, είναι, κατανόητο το να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ε, αλλά είναι θέμα αρμοδιοτήτων. Και εγώ ίδιο δεν ξέρω τι να πω, διότι από τη μία καταλαβαίνω του αναφέροντε, από την άλλη καταλαβαίνω και τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, Ρόζα. Εγώ ήθελα απλώ να επιθυμήσω το εξή ε, ε, ε, συζητήσαμε και με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και είπε ακριβώ αυτό που είπε ο Πίτερ, ότι δεν είμαστε αρμόδιοι. Κοιτάξτε, ε, εγώ θα ακολουθήσω αυτό που θα πείτε, αλλά ε, κοιτάξτε, εάν δημιουργούμε προσδοκίες οι οποίες δεν μπορούν να οδηγήσουν πουθενά, δεν έχει και πολλή έννοια. έχετε το λόγο ξανά. Ε, κοιτάξτε, εγώ επιμένω. Η Επιτροπή διαρκώς λέει ότι δεν είμαστε αρμόδιοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Μπορεί να προσπαθήσει, μπορεί να συνεχίσει και να προσπαθεί να πιέζει την Κομισιόν έτσι ώστε να πάρει πολιτικές αποφάσεις που θα λύσουν τέτοια κατάσταση. Έχει και πόρους, ε, η Κομισιόν έχει πόρους και μπορεί να το κάνει κατά την άποψή μου. Επανέρχομαι και επαναλαμβάνω και επιμένω. Έχει διπλή γλώσσα. Αυτή η διγλωσσία. Ε, τι κάνει. Στην ουσία πετάει την μπάλα στην κερκίδα, στην εξέδρα. Για να το πω έτσι πολύ απλά και ποδοσφαιρικά. Και ε, ε, τι να σας πω σε σχέση με αυτά που είπατε για την ε, τοπική κυβέρνηση της Γαλλικίας και την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας ε, δεν νομίζω πια ότι κάνανε και τόσα πολλά πράγματα γιατί ακόμα βρισκόμαστε εδώ έχουμε απέναντί μας ε, την, τον σύλλογο των μεταναστών που έχουν επιστρέψει στη Γαλλικία και είναι συνταξιούχοι και έχουν τέτοια προβλήματα κάτι δεν έγινε και τόσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πράγματα. Πρώτον, ε, η Οικονομική Επιτροπή αυτό που είπε είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν ε, να ακολουθήσουν την δικαστική οδό για να επιτύχουν τα δικαιώματά τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό το ξέρουμε, βρίσκεται και γραμμένο στις συνθήκες. Δεύτερον, ναι, όντως έχει υπάρξει διακριτική μεταχείριση. Π.χ. Ε, ένας Ισπανός που ας πούμε από την κυβέρνηση της Ισπανίας παίρνει δύο συντάξεις, ε, μία κανονική και μία αναπηρίας, ε, θεωρείται ότι παίρνει μία σύνταξη. Εάν αυτός ο συγκεκριμένος πάει στην Ισπανία και παίρνει μία σύνταξη ε, γύρατος ας πούμε ε, από την Ισπανία και άλλη μία από την ε, Γαλλία το ίδιο θα θεωρήσει μία σύνταξη. Δεν είναι δυνατόν όμως να θεωρήσει η Ισπανία δεύτερον, δεύτερον πληρωτή κάποιος, κάποιον ο οποίος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το ζήτημα της αναπηρίας είναι παράνομο είναι παράλογο, συγγνώμη, να μην αναγνωρίζεται η αναπηρία σε έναν εργαζόμενο, αναπηρία 100% ε, ε, που έχει αναγνωριστεί η αναπηρία του σε μία χώρα ε, και δεν είναι δυνατόν η Ισπανία να μην αναγνωρίζει την αναπηρία αυτή όταν αυτός ο άνθρωπος μεταναστεύσει ξανά στην Ισπανία ε, δεν, δεν, ε, ε, εδώ υπάρξει, υπάρχει μια ε, ε, διαστροφή ας πούμε των αρχών κάποιος ε, που έχει αναγνωριστεί ως ανάπηρος στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεται ως τέτοιος ε, στην ε, Ισπανία. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όποιες διεκδικήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, γιατί απαιτούνται από την ισπανική πλευρά λεπτομερέστατα έγγραφα από την αρχή της άλλης χώρας, η οποία αποφάσισε αποφάσισε και αναγνώρισε την αναπηρία. Επομένως, εμείς ζητούμε, εάν έχει αναγνωριστεί ε, η αναπηρία σε μία χώρα μέλος, αυτή η αναπηρία να αναγνωρίζεται και σε μια άλλη χώρα. Κυρίως δε αν έχει δοθεί και σύνταξη στον ε, ανάπηρο, γιατί διαφορετικά όλες οι εργασίες και οι προσπάθειες είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Ε, κατά τα άλλα, ναι, ε, προκύπτει ε, φορολογική απέτηση λόγω της προέλευσης των συντάξεων. Τέλος, ε, πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς δεν έκανε τίποτα η τοπική κυβέρνηση της ε, Γαλλικίας απέναντι στην κατάσταση και απέναντι στους εκπροσώπους των, και τις οργανώσεις των συνταξιούχων. Ε, στην ουσία αυτό που κάνει η Ισπανική κυβέρνηση είναι να εφαρμόζει ε, με αναδρομική ισχύ ε, κάποιες φορολογικές επιραβαρήσεις σε συντάξεις πηγαίνοντας και τέσσερα χρόνια πίσω. Εάν η Ισπανική κυβέρνηση αλλάξει κριτήρια και εάν ε, αρχίσει να ε, απαιτεί ε, αλλαγές και να απαιτεί πληρωμές από ξένους και αρχίζει να έχει αυτή η απέτηση και αναδρομική ισχύ, τότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση, κυρίως δε για ανθρώπους που όπως είπα και προηγουμένως ζουν στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση έχει ως εξής. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την Επιτροπή Αναφορών, διότι έτσι μπορούμε να έχουμε άμεσο διάλογο πάνω σε προβλήματα. Από την άλλη, κύριε Πορτέλα, με όλη τη συμπάθεια που σας τρέφω, είχαμε τη δυνατότητα να υπερψηφίσουμε αυτήν, πάνω σε αυτήν την συνεχιζόμενη διάκριση. Θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε και να και να υπερψηφίσουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε διάφορες ε, συνθήκες, ε, συμφωνίες, ε, υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές που απορρέουν από τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Εγώ προτείνω το εξή. Να γράψουμε τρεις επιστολές στο όνομα της Επιτροπής Αναφορών. Να στείλουμε μία επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση, στην οποία να την ενημερώνουμε σχετικά με την ύπαρξη αυτού του προβλήματος. και να προτείνουμε λύση ενδεχομένως αναδρομική που να ε, συνάδει με την πρότασή σας. Ταυτόχρονα να στείλουμε επιστολή στην τάξου, στη Διεύθυνση Τάξου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου να τους ενημερώνουμε σχετικά με το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ένα απομονωμένο διμερές πρόβλημα, είναι πρόβλημα που απαντάται και σε άλλες περιπτώσεις, ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία, για παράδειγμα. Επίσης, καταλαβαίνω ότι το θέμα της εναρμόνισης της φορολογίας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και ότι δεν θα δούμε σύντομα επίλυση του προβλήματος. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, Ίσως να μπορέσουμε σύντομα να έχουμε κάποια λύση. Και να στείλουμε επιστολή στην Επιτροπή ΕΚΟΝ να λέμε ότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα αυτό και να τους ζητάμε να βρουν λύση. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, κύριε Πόρτελα, δυστυχώ δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε αυτέ τι τρει επιστολέ και να κλείσουμε την ε, αναφορά. Η κυρία Στανόκα. Νομίζω, νομίζω ότι για το θέμα της αναπηρίας και των συντάξεων αναπηρίας να απευθυνθούμε και στην Επιτροπή Απασχόλησης για την αρμόδια. Συμφωνώ. Α το πράξουμε αυτό. Εγώ θα πρότεινα να σταλεί νέα επιστολή στο Συμβούλιο από τη στιγμή που μιλούμε για τα κράτη-μέλη λοιπόν και να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά τουλάχιστον μέχρι να απαντήσει το Συμβούλιο. Κανένα πρόβλημα με αυτές τις αλλαγές δέχομαι την πρόταση θα κλείσουμε την αναφορά λοιπόν μετά από όλα αυτά τα βήματα. Συμφωνείτε? Καλώς. Εγώ νομίζω ότι στην επιστολή που θα στείλουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης, εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση, να τους ζητήσουμε να μελετήσουν την εναρμόνιση. δηλαδή να ξεκινήσουν τη μελέτη αυτού του θέματος προκειμένου να καταφέρουν την εναρμόνιση κάποια στιγμή. Είναι πρότασή μου αυτή. Κανένα πρόβλημα και αυτό είναι αποδεκτό. Έτσι λοιπόν θα χειριστούμε αυτό το ζήτημα σήμερα. Αυτά λοιπόν για αυτό το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω. Καλή σας όρεξη. Θα τα πούμε στις 3.